που δεν υπάρχουν θεωρούμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Και τώρα θα πρέπει να σα ενημερώσω ότι αύριο ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και εγώ πρόκειται να υπογράψουμε κάποιε νομοθετικέ πράξει δυνάμει τη ε, συναπόφαση ε, βάσει τη διαδικασία 74 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι δε τίτλοι αυτών των ε, πράξεων πρόκειται να μνημονηθούν ή στα πρακτικά.